η συζήτηση για το θέμα αυτό. Όχι μόνο η συζήτηση, αλλά κλείνει και η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Αφού σας πω όμως ότι η